Σύνοδος. Καταρχάς, ε, μία ανακοίνωση έχουμε να σας κάνω. Χτες στη Σαουδική Αραβία 7 εκτελέστηκαν. Είναι πραγματικά λυπηρό ότι οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας αγνοούν τις ε, ενστάσεις ε, της διεθνούς κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατάργηση της